αντίρρηση. Συνεπώς, έληξε η συνεδρίαση. αυτή. Τα πρακτικά θα ε, τεθούν προς ε, έγκριση στην αρχή της ε, επόμενης συνεδρίασής μας, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Οι αποφάσεις οι σημερινές θα υποβληθούν στους αποδέκτες τους και στις αρμόδιες αρχές. Λίγη συνεδρίαση αυτή. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Καλή σας όρεξη.